Συνεχίζουμε στο επόμενο θέμα. Έχουμε τέσσερα σχέδια ψηφίσματος για το Λάος και το Βιετνάμ και θα ήθελα να δώσω το λόγο στους ε, συντάκτες της, ε, των ψηφισμάτων, ε, μεταξύ άλλων στην κυρία Ντεκάιζερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχουμε ένα νέο κατεπήγον για το Λάος και το Βιετνάμ. Δεν είναι πρώτη φορά που έχουμε το θέμα αυτό κατεπήγον στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά αυτό το ψήφισμα τουλάχιστον δεν θα πρέπει να μείνει κενό γράμμα. Ανησυχούμε σοβαρά, γιατί από το 2006 ε, το Βιετνάμ ε, εξήλθε από τον κατάλογο της Ηνωμένων Πολιτειών για την καταστολή και την καταστρατήγηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Παρ' όλα αυτά εξακολουθεί η κυβέρνηση να καταπιέζει τους αντιφρονούντες. Εγώ θα αναφερθώ στην κυρία Τρανξ τι που έχει blogger, είναι δημοσιογράφος, είναι ακτιβίστρια και βρίσκεται στη φυλακή για πολύ αμφίβολους λόγους. Το πιο πιθανό είναι να βρίσκεται γιατί εκφράζει ελεύθερα τη γνώμη της και προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Υποφέρει από διαβήτη, είναι φυλάσθενη και έχουμε σοβαρούς ε, φόβους για την υγεία της. Ε, δεν ζητούμε μόνο τη χαλάρωση των συνθηκών φυλάκισης, αλλά την άμεση απελευθέρωσή της. Μας ενδιαφέρει το Βιετνάμ, είναι μια μεγάλη χώρα και μάλιστα θα αναλάβει την Προεδρία του ΑΣΕΑΝ το 2010 και πιστεύω ότι η θέσπιση μέτρων που θα συνάδουν με τους διεθνείς κανόνες της δημοκρατίας ε, είναι κάτι που θα ενισχύσει το ηθικό κύρος αυτής της χώρας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Στόμεσμαν. Έχει το λόγο για δύο λεπτά. Η κατάσταση για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Βιετνάμ είναι ενισχυτική. Θρησκευτική δίωξη χριστιανών και βουδιστών ιδίω είναι καθημερινό φαινόμενο. Όποιο προσπίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα ελέγχεται συστηματικά. Το Σεπτέμβριο εκατοντάδες ε, ε, μοναχών ε, έδιχαν επιθέσεις, αρχή. η αστυνομία αδρανούσε εκείνοι που είχαν πάει στο ναό που ακούει ε, έτυχαν ε, επιθέσεων απαραδέκτων. Εμείς ε, θα πρέπει και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από άλλες μεριές του κόσμου να προασπίσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μέχρι τώρα δεν έχουμε εισακωστεί. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι του χρόνου το Βιετνάμ θα αναλάβει την Προεδρία της Ομάδας Κρατών ΑΣΙΑΝ. Στο Λάζ δεν είναι καλύτερη κατάσταση. Αρχές Νοεμβρίου πάνω από 300 ελληνικοί διαδηλωτέ που ζητούσαν περισσότερο πλουραλισμό και δημοκρατία ε, δάχθηκαν άγρια από την μυστική αστυνομία. Οποιοδήποτε πολιτικός διάλογος στη χώρα αυτή καταστρέφεται εκ μιας αρχής από την, το ενιαίο κρατικό ε, κόμμα το ίδιο ισχύει για τις 5.000 ε, προσφύγων Λαομόν που αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε στρατόπεδα στην Καμπότζη. Δεν τους ε, δίνεται όμως το καθεστώς ε, του πρόσφυγα. Η οργάνωση για τρίχωρη Σύνορα που ήταν και εδώ είχε μια παρουσίαση στο Κοινοβούλιο είπε ότι δεν μπορεί να προσφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στους ανθρώπους αυτούς γιατί συνεχώς συλλαμβάνονται κάποιοι άνθρωποι και τους υποχρεώνουν να επιστρέψουν στο λαός και λέγεται ότι το κάνουν ε, ε, ακούσια, αλλά αυτό, εκούσια, αλλά αυτό δεν είναι, δεν είναι σωστό. Υπάρχουν συμφωνίες και με τις δύο χώρες αυτές όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και δημοκρατία. Τι πραγματοποιήθηκε από αυτά. Πρέπει να τους ρωτήσουμε και θα πρέπει να ασκηθεί πίεση στις κυβερνήσεις του Βιετνάμ και του Λάος. Ευχαριστώ. Arvoisa puhemies, on Σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι είναι πολύ καλή είδηση ότι τα κράτη του ΑΣΕΑΝ δημιούργησαν ένα περιφερειακό θεσμικό όργανο για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό είναι και πολύ λογικό και πολύ σημαντικό. Να έχουμε επαφές με τους ε, ε, βουδιστές μοναχούς που υπέστησαν ε, διώξεις και κακοποίηση. Νομίζω ότι θα πρέπει να ζητήσουμε επίμονα σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Βιετνάμ και να καταδικάσουμε το γεγονός ότι πάνω από 300 μοναχοί άνδρες και γυναίκες σε διάφορα μοναστήρια κακοποιήθηκαν. πολύ πιστοί διώκονται στο Βιετνάμ και στο Λάος. Γι' αυτό ζητούμε στο ψήφισμα ο ειδικό εκπρόσωπος του ΟΗΕ που ασχολείται με την ελευθερία θρησκευτικής πίστης να επιληφθεί ε, του θέματος. Εκ μέρους του ΕΛΚ το λόγο έχει ο κύριος Κριστιαν Πρέντα για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ. călugărilor buditi survenit la lui septembrie cred eu faptul că vietnamul refuză să drepturilor omului. Ό,τι δεν να τα δικαιώματα. στο ότι οι των διαδηλώσεων των εξακολουθούν να κρατούνται Όποια προσπάθειε έγιναν για την πρόσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων καταστάλησαν άκρια και όσοι συμμετείχαν στι διαδηλώσει αυτέ διώχθησαν. Αυτέ οι δύο χώρε πρέπει όμω να σεβαστούν το διεθνέ δίκαιο για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η προστασία των μειονοτήτων, η προστασία εκείνων που προσπαθούν να ε, ασκήσουν τα θρησκευτικά του δικαιώματα πρέπει να τύχει σεβασμό. Θα πρέπει να παρακολουθήσουμε στενά την, κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις χώρες αυτές και να δράσουμε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κυρία Γκέριγκερ Ντεόντεμπερ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Η συνέχιση των διαπραγματεύσεων για τη νέα συμφωνία συνεργασίας και εταιρική σχέσης με το Βιετνάμ θα πρέπει να περιλαμβάνει και για τα ανθρώπινα δικαιώματα, γιατί από τις πληροφορίες μας μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η κατάσταση είναι πολύ ανησυχητική, καταπιέζονται και διώκονται ακόμη και άνθρωποι που έχουν blogger στο ίντερνετ. Είναι πολύ ανησυχητική η κατάσταση. Μάλιστα, ε, οι διατάξεις του Βιετνάμ για τη χρήση του διαδικτύου περιορίζουν την ελευθερία έκφρασης, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δημοκρατικά δικαιώματα. Θα επίσης, περιορίζεται ακόμη και η πρόσβαση Μπορείτε να επιβραδύνετε λίγο κυρία Γκέριγκερ γιατί δεν μπορώ να σας προλάβουν οι διερμηνείς. Προσπαθώ, κάνω την μπορώ, αλλά σε ένα λεπτό τι να πρώτο προλάβω. Ε, το 2008 οι διατάξεις για τα μπλοκ ε, περιλα... περιορίζουν όχι μόνο τα προσωπικά δικαιώματα, αλλά και την ελευθερία τύπου και μάλιστα έχουν, ε, ορισμένοι μπλόγκερ έχουν καταδικαστεί για υποδαβλισμό αντικυβερνητικών ενεργειών και προσπάθεια υπονόμευση τη κυβέρνηση. Δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην είναι διάφορη για αυτά τα ανησυχητικά φαινόμενα στο Βιετνάμ. Και εκτό από τα πολιτικά διαβήματα θα πρέπει να γίνουν κάποια νομικά διαβήματα. Γι' αυτό απευθύνω έκκληση στη νέα συμφωνία εταιρική σχέση και συνεργασία με το Βιετνάμ, οπωσδήποτε να συμπεριλάβουμε και ερήτερα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σα ευχαριστώ, κύριο Βαμπάλεν, εκ μέρου των Φιλελευθέρων. Οι φιλελεύθεροι θεωρούν ότι το Λάος και το Βιετνάμ δεν είναι δημοκρατικές χώρες. Δεν υπάρχουν εγγυήσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ούτε και για τα θρησκευτικά σε καμία από τις δύο χώρες. Γι' αυτό και υποστηρίζουμε το ψήφισμα αυτό και ζητάμε από το Συμβούλιο να πάρουν τα κατάλληλα μέτρα. I thank you very much. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα και εγώ να υπογραμμίσω την ε, δραματική κατάσταση ε, που ζουν οι χριστιανοί στο Βιετνάμ. Εξαιτίας ε, της κυβερνητικής τάση. υπήρξαν καταπιέσεις, διώξεις, βανδαλισμοί σε μοναστήρια, κατά, κατά καθολικών και προτεστάντων ιερέων. Οι η χριστιανική θρησκεία θεωρείται ως θρησκεία που εξυπηρετεί υπεριαλιστικά συμφέροντα στο Βιετνάμ. Οι καταπιέσεις είναι πολλών μορφών, φυλακίσεις, βασανιστήρια, περιορισμοί κατοίκων, εγκλισμοί σε ψυχιατρικά ιδρύματα. Τέτοιες πρακτικές δεν μπορούν να αφήσουν αδιάφορη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει οπωσδήποτε να λάβουμε κάποια μέτρα. Δεν μπορούμε να γινόμαστε μάρτυρες τέτοιας καταπίεσης ε, πιστών της χριστιανικής θρησκείας. Γιατί πραγματικά είναι βάρβαρη η στάση που κρατάει το Βιετνάμ απέναντι στους πιστούς ε, χριστιανούς. Σας ευχαριστούμε κύριε Λεγκούτκο. Η κυρία Κορχόλα, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Κάναμε ένα πολύ σημαντικό... Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το Λάος έκανε ένα πολύ σημαντικό βήμα το μήνα Σεπτέμβριο, βελτιώνοντας την κατάσταση. Σε ό,τι αφορά την ελευθερία της έκφρασης ε, και πολιτικής σκέψης. Αυτά όμως στη θεωρία, γιατί στην πράξη ελάχιστη πρόοδος έχει σημειωθεί. Και από τα λόγια μέχρι τα έργα υπάρχει τεράστια απόσταση μερικές φορές. Εμείς θα πρέπει να γεφυρώσουμε αυτό το κενό. Στη, διαδικασία του, στη δεκαετία του 90 έγιναν πολύ σημαντικές διαμαρτυρίες και διαδηλώσεις και εκατοντάδες φοιτητέ συνελήθησαν. Το ίδιο συνέβη και στις ειρηνικές διαδηλώσεις του προηγούμενου Μαρτίου. Η κυβέρνηση, και οι αρμόδιες αρχές λένε ότι θέλουν να βελτιώσουν την κατάσταση και να υιοθετήσουν κάποιες νομοθετικές μεταρρυθμίσεις το συντομότερο δυνατό. Οι νέε όμω νομοθετικέ ρυθμίσει θα πρέπει να συνάδουν με το διεθνέ δίκαιο, γιατί το Λάο έχει αναλάβει δεσμεύσει ε, να εγκρίνει νομοθεσία που θα ακολουθεί το διεθνέ δίκαιο. Θα πρέπει το Λάο να γίνει μια ε, δημοκρατία με την πραγματική σημασία του όρου. Ο Μάρκ Ταραμπέλα για ένα λεπτό. Πράγματι το 2009 ήταν μια χρονιά κατά τη διάρκεια της οποίας το Βιετνάμ έκανε κάποια βήματα ανοίγματο. ή μάλλον αυτό έγινε πριν δύο χρόνια. Δεν ήταν ικανοποιητικά όμως αυτά τα βήματα και συνεχίζεται η καταστολή των θρησκευτικών δικαιωμάτων όπως και οι συλλήψεις ε, μοναχών βουδιστικής ε, καταγωγής. Πιστεύουμε μέσω του ψηφίσματος αυτού λοιπόν να θυμίσουμε τη σημασία που έχουν τα ανθρώπινα δικαιώματα μιας και πρόκειται να αναλάβει και την Προεδρία του ΑΣΕΑΝ. Έχει επίσης επικυρώσει την διεθνή, το Διεθνές Σύμφωνο για τα πολιτικά και θεμελιώδη δικαιώματα και θα πρέπει να γίνει πλήρης σεβαστή η υπογραφή του στον τομέα των προσωπικών δικαιωμάτων. Και επίσης θα πρέπει να απελευθερωθούν όσοι συνελήφθηκαν στις 2 Σεπτεμβρίου του 2009, όπως και οι φυλακισμένοι από το 1999. Τσαρνιέσκι. Ευχαριστώ. Εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μίλησαμε για το Βιετνάμ ε, μιλώντας για την ε, θρησκευτική δίωξη που υπέστησαν ε, οι βουδιστές. Αυτό έγινε στην προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία. Σήμερα μιλούμε πάλι για την παραβίαση των θρησκευτικών δικαιωμάτων και στις δύο χώρες, και στο Βιετνάμ και στο Λάος, αλλά εδώ θύματα και διωκόμενοι είναι χριστιανοί. Λυπούμε που η δίωξη πιστών έχει γίνει πραγματικότητα και καθημερινότητα στις δύο αυτές χώρες. Καμία, κανένα σεβασμός ούτε για τις θρησκευτικές μειονότητες ούτε για τις μειονότητες εν γέννη. Δεν μπορούμε να μείνουμε διάφοροι. Ε, θα ήθελα να μιλήσω ως blogger και γνωστός blogger στην Πολωνία να εκφράσω τη διαμαρτυρία μου έναντι των διώξεων αυτών κατά των συναδέλφων blogger στο Βιετνάμ. Νομίζω ότι θα πρέπει να υψώσουμε τη φωνή μας υποστηρίζοντας τους μπλόγκερ στο Βιετνάμ. Σας ευχαριστώ τώρα διαδικασία του Catch the Eye. Ο κύριος Μάουρο για ένα λεπτό. Διώξεις, διακρίσεις επιθρησκευτικής βάσεως. Αυτό δεν είναι κάτι το καινούριο στο Βιετνάμ. Κρατάνε εδώ και 50 χρόνια. Τα πιο πρόσφατα επεισόδια είναι η επιδρομή της αστυνομίας στην, στον καθεδρικό του Λόγκ που σταμάτησε να λειτουργεί σαν εκκλησία και έγινε δημόσιο πάρκο όπως επίσης και η καταστροφή του νεκροταφείου του καθολικού του Χανόη και μάλιστα όχι μόνο είναι θύματα οι χριστιανοί αλλά δικάζονται πολλές φορές και κατηγορούνται σαν εγκληματίες για λόγους πίστης. και μάλιστα έχουν μπλοκαριστεί και ε, τρεις ε, ιστοτόποι στο διαδίκτυο στο Βιετνάμ που κυκλοφορούν ε, ενημερωτικά στοιχεία για τις κινήσεις των διοκτικών αρχών. Καταδικάζονται οι χωρικοί που έχουν χριστιανική πίστη ότι είναι πολύ συχνά ε, υπόλογοι ποινικά για διάφορα εγκλήματα κτλ. Νομίζω ότι η συζήτηση αυτή είναι πολύ εύθετη για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα πρέπει τα ανθρώπινα δικαιώματα να προστατεύονται παντού στον κόσμο, λέει ο κύριος Ζόμπρο. Όταν συζητάμε βέβαια για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις που έχουμε μπροστά μας τώρα θα πρέπει να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί ιδιαίτερα στις χώρες όπου παραβιάζονται μαζί με τα πολιτικά δικαιώματα και τα θρησκευτικά αντίστοιχα. Θα πρέπει να προστατεύουμε τα θρησκευτικά δικαιώματα και ο καθένας θα πρέπει να είναι ελεύθερος να πιστεύει αυτό το οποίο επιλέγει. Τέτοιες περιπτώσεις λοιπόν πρέπει πάντα να έρχονται στην επικαιρότητα και να καταδικάζονται. Εμείς βέβαια στην Ευρώπη γεωγραφικά βρισκόμαστε πάνω σε μια ήπειρο η οποία δεν αντιμετωπίζει τέτοια προβλήματα θεωρητικά και θα πρέπει να είναι το παράδειγμα για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Φυσικά και υπάρχουν προβλήματα όμως και σε μας. Δεν υπάρχει βέβαια σύγκριση στη σοβαρότητα των προβλημάτων. Ανησυχώ όμως για την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με την ανάρτηση του θρησκευτικού συμβόλου στην Ιταλία. Νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό προηγούμενο. Κλείνοντας, λέει ο κύριος Ζόμπρο. Πάντα υπερασπιστήκαμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Ευχαριστώ. Charles Τάνοκ, ο τελευταίος ομιλητής. Δυστυχώς το Βιετνάμ και το Λάος μαζί με την Κούβα και τη λαϊκή δημοκρατία της Κίνας παραμένουν μονοκομματικές κομμουνιστικές δημοκρατίες. Ενώ η ελευθερία του τύπου, η δημοκρατία, ελεύθερες εκλογές και η ελεύθερη άσκηση θρησκευτικών δικαιωμάτων έχουν κυριαρχήσει σε πάρα πολλές περιοχές του κόσμου στο Βιετνάμ διώκονται οι Βουδιστές και όχι μόνο και επίσης διώκονται η μειονότητα των χμόγ στην λαϊκή δημοκρατία του Λάος. Θα πρέπει λοιπόν να ανταλάβουμε υπόψη μας αυτά και οι κομμουνιστικές δημοκρατίες ποτέ δεν θα λειτουργήσουν από μόνες τους σαν ελεύθερες δημοκρατίες. Επίτροπος Δεχούχτ. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα σας μιλήσω πρώτα για το Λάος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι τα τελευταία χρόνια υπήρξε μια αισθητή βελτίωση στην πολιτική κατάσταση στο Λάος και συμφωνεί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι η επικύρωση από το Λάος τη, της Διεθνούς Συμφωνίας για τα πολιτικά, και, για τα πολιτικά δικαιώματα είναι σημαντικό, βήμα πρόοδου που κατοχυρώνει την ελευθερία της, του τύπου, του, της έκφρασης, του συνεταιρίστε κλπ. Επίσης υπέγραψε και το, τη Διεθνή Σύμβαση κατά της διαφθοράς. Επίσης έχει εγκρίνει ένα νόμο για την αναγνώριση των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Είναι σημαντικός ο ρόλος τους σε μια δημοκρατική κοινωνία και στην δημοκρατική ανάπτυξη μιας χώρας. Σε ό,τι αφορά τους πολιτικούς κρατουμένους, σε ό,τι αφορά τους τρεις ανθρώπους που επισημάνατε, οι αρχές ε, τον Οκτώβριο του 2009 δήλωσαν σε μια αντιπροσωπεία στην Κενσιάνο ότι ο κύριος Γκέτσια ήδη απελευθερώθηκε, ήδη απελευθερωθεί από το 2002. Δύο από τους, άλλους, από τους τρεις, ο κύριος Εγκαλούγκ Φινγκφάν και ο κύριος Τόγκ Πασέντ και Κόγκ αναφέρεται ότι χαίρουν άκρας υγείας και η κυβέρνηση δεν γνωρίζει τίποτα για τον κύριο Μπουβάν Σαν Μανιβάν. Δεν ευθύνομαι καθόλου για την προφορά μου, λέει ο Επίτροπος. Μάλιστα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, συζήτησε με πρεσβευτές ε, για να διευκρινίσει κατά πόσο ευσταθούν οι ισχυρισμοί για τις συλλήψεις 300 ατόμων τον Νοέμβριο του 2009 μετά από διαδήλωση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφωνεί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι η κράτηση 158 ατόμων στο Νούνκαϊ χρήζει άμεσης λύσης και μάλιστα ζητεί από τις κυβερνήσεις του Λάους και της Ταϊλάνδης να επιτρέψει τους φυλακισμένους, κρατουμένους να εγκατασταθούν σε τρίτες χώρες που προσέφεραν άσυλο σε ό,τι αφορά τη, τα στρατόπεδα κράτησης λατιανών χμόγκ στην Ταϊλάνδη θα πρέπει να το εξετάσουμε. Για το Βιετνάμ τώρα. Συμμεριζόμαστε τις ανησυχίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για πρόσφατε ενδείξεις σκληρής τάσης του Βιετνάμ σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και σε ό,τι αφορά οι πρόσφατε ε, συλλήψεις ε, φιλιρινικών blogger ε, ή διαδηλωτών οι μοναχών από τη βουδιστική κοινότητα δημιουργούν πραγματικά σοβαρές ανησυχίες για την κατάσταση στο Βιετνάμ στην Ευρώπη. Απευθύνουμε έκκληση στο Βιετνάμ που είναι μέλος του Μηχανισμού Οικουμενικής Περιοδικής Επανεξέτασης ε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα να απελευθερώσει όλους τους πολιτικούς κρατουμένους και ιδιαίτερα το Λί Τίν, συγγραφέα και εκτιβίστρια θεμελιωδών Θεμελιών Δικαιωμάτων και τον ιερέα Χιου Βαγγλή που κρατείται αυτή τη στιγμή επειδή απλώς φιλιρινικά εξέφρασε τις απόψεις του. Ε, πιο ανεξάρτητα μέσα μαζικής ενημέρωσης θα μπορούσαν να διδραματίσουν σημαντικό ρόλο στον εκδημοκρατισμό του Βιετνάμ. Θα ενθαρρύνουμε τη χώρα αυτή να υιοθετήσει νομοθεσία για τον τύπο που θα συμφωνεί με τις διεθνείς συμφωνίες για την ελευθερία τύπου. Θέλουμε έναν όριμο ε, διάλογο ανθρωπίνων δικαιωμάτων με το Βιετνάμ και περιμένουμε τις δεσμεύσεις αυτής της χώρας και την έμπρακτη εφαρμογή τους. Και για να προχωρήσουν οι συμφωνίες μας ε, και ο διάλογος θα πρέπει να δείξει αυτά σημάδια εφαρμογή των δεσμεύσεων του Βιετνάμ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Έχει τελειώσει η συζήτηση για το θέμα αυτό και έχουμε τελειώσει το ζήτημα αυτό για το Λάος και το Βιετνάμ. Ακολουθεί η συζήτηση σχετικά με πέντε ψηφίσματα για την Κίνα, μειωνοτικά δικαιώματα και θανατική ποινή. Δίνω καταρχήν το λόγο στην κυρία Ντεκέζε. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η ομάδα μου έχει αποσύρει την